Ε, εκπρόσωποι της Κομισιόν, συνεργάτες. Είναι η τελευταία ευθεία πριν από τις διακοπές. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ε, έχουμε λοιπόν... Έχουμε την υπόθεση ε, του εξυγχρονισμού των τελενίων με μια επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας την προηγούμενη εβδομάδα και μια ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση Ριβαλίνη για το δεύτερο σχέδιο απαλλαγής για το Συμβούλιο. Οι συντονιστές είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν την Προεδρία του Συμβουλίου και ο κύριος Ριβελίνη φαντάζομαι ότι θα καταγράψει στην έκθεση του τα συμπεράσματα από την εν λόγω συνάντηση. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θα περάσω στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Και ως συγητής έχω να σας παρουσιάσω την γνωμοδότησή μου για την εξυγχρονισμό των τελωνιακών υπηρεσιών. Ε, όπως γνωρίζετε έχω κάνει μια γνωμοδότηση την έχω καταθέσει. Προσπαθώ στο να είναι πιο σύντομη και στο περιεχόμενο και στην έκθεση. Προσπαθώ να περιγράψω την, ε, τα δεδομένα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, ξελίσσονται αυτοί οι τελωνιακοί έλεγχοι. Ασφαλώς αποτελεσματικοί ε, τελωνιακοί έλεγχοι αποτελούν πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν βέβαια σημαντικούς πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ε, πόροι αποδασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ε, φυσικά πέραν των δασμών η τελωνιακή έλεγχη ε, συμβάλλουν στην αποτελεσματική ίσπραξη του ΦΠΑ και την καταπολέμηση της ε, απόπειρας διαφυγής καταβολής του φόρου θέμενες αξίες. Μιλάμε λοιπόν για 16 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα άμεσα από τελωνιακούς δασμούς και έμεσα από την ίσπραξη ΦΠΑ χάρη στα τελωνία μέσα σε ένα έτος μόνο για το 2011 συγκεκριμένα. Όταν δε, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά τα τελωνία μας, ε, αυτό έχει επιπτώσεις ορατές αμέσως στις επιχειρήσεις μας, γιατί πέφτουν αυτές θύματα της διαφυγής του ΦΠΑ, των ε, άλλων ε, ανταγωνιστών. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι είχαμε θεσπίσει μια ειδική επιτροπή, ερευνητική επιτροπή που ασχολήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την απάτη σε επίπεδο τελωνίων, τελωνιακή απάτη, την ε, δάσμο διαφυγή και πολλοί είχαν διερωτηθεί το επίπεδο ε, των όρων που έχουν ε, να εφαρμόσουν τα τελωνία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν είναι ισοδύναμο, αν υπάρχει αυτό που λέμε στα αγγλικά level playing field, εάν υπάρχει ε, ανάγκη και πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των αρχών αυτών των τελωνιακών που να λειτουργεί γρήγορα, στιγμιαία θα λέγαμε και με πληρότητα. Και για να προχωρήσω, επισημαίνω ότι έχουμε συμπεριλάβει, ύστερα από μια ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το, την απλούστευση των διαδικασιών σε τελωνιακό επίπεδο, μια πρόταση, μια παράγραφο στην ε, γνωμοδότησή μου, με στόχο οι τελωνιακές διατυπώσεις ε, να περιοριστούν στο ελάχιστο αποδεκτό. Με βέβαια σωστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Δεν πρέπει να λησμονούμε όμως ότι το 70% μερίδα του λέοντος δηλαδή όλων των διαδικασιών ε, μπορεί να εντάσσονται σε αυτήν την ε, Είχαμε πάρα πολλές απώλειες εσόδων με πολλές απάτες και διαφυγή ε, καταβολής δασμών ε, σε επίπεδο τελωνίων. Και γι' αυτό σημειώνω στην επόμενη παριθμόν 5 παράγραφο ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα συστημικό ε, ένα συστημικό έλεγχο, δηλαδή να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ελέγχου, ακόμα και σε περίπτωση απλουστευμένης τελωνιακή διαδικασία, επαρκή και εκ των υστέρων έλεγχος, που βέβαια θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, όπως άλλωστε είχε και στο παρελθόν υπογραμμίσει το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο είχε ζητήσει επισταμένως η ανάλυση του κινδύνου να εκτελείται με βάση μια αυτόματη ανάλυση δεδομένων την εποχή εκείνη είχε καταγγείλει το ελεγκτικό συνέδριο, ήταν λίγα τα κράτη εκείνα που ακολουθούσαν αυτή την πρακτική και πρέπει να στήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει για την γενίκευση της ε, διαδικασίας αυτής. Το δε έβδομο σημείο, ξέρετε ότι δεν θα μπορούσα ούτως ώρες να ομολογήσω να περιλάβω οτιδήποτε θα ήθελα στο κείμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνουμε στο σημείο 7 παραπομπή στην απαλλαγή στο ψήφισμα της 10 Μαΐου του 2011, το κείμενο εκείνο του κυρίου Χατζημαρκάκη και το ψήφισμα που περιλαμβάνει όλες τις ειδικές εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και στο τρίτο τμήμα του ψηφίσματος αυτού. Θα θυμάστε ότι είχαμε περιλάβει ένα ειδικό κεφάλαιο για τα τελωνία και τις ερωνιακές διατυπώσεις και έτσι πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να ε, συμφωνήσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα μπορούμε να τα διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Αυτή ήταν η γνωμοδότηση. Ελπίζω να έχετε κάποιες παρατηρήσει. Πολύ φορές θα τις ακούσω ε, για να τις ενσωματώσω στο κείμενό μου. Κύριο Σίταλα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται εδώ ε, για μια εξαιρετική αρχή, μια εξαιρετική βάση για την περαιτέρω εργασία μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Γνωρίζω λίγο το τελωνιακό σύστημα συνήθως ε, ε, στα όσα συμβαίνουν ε, στα σύνορα της χώρας μου με την Ρωσία. Γνωρίζω λοιπόν και τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα σύνορα με μια τρίτη χώρα. Η αυτόματη μετάδοση δεδομένων ε, ε, είναι κάτι που μας ε, χρειάζεται απόλυτα και επίσης η ανάλυση κινδύνου είναι, έχει μεγάλη σημασία. Η Επιτροπή φέρεται σαν να υπάρχει μονάχα μία τελωνιακή υπηρεσία και λες και το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, όμως χρειαζόμαστε πραγματική εναρμόνιση ε, και επικαιροποίηση των συστημάτων μας, διότι η παρούσα κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, είναι, ε, πρέπει πάντως να παραδεχτώ ότι είναι πάρα πολύ καλές οι προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Τζουρίμπιχ έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ένα ερώτημα το οποίο επανέρχεται. Ποια είναι η σύγκριση μεταξύ των απατών για το ΦΠΑ και των απατών για, τα, για τους τελωνιακούς δασμούς. Έχουμε στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε μια επακριβέστερη εικόνα για τις τελωνιακές απάτες. Άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλαν να λάβουν το λόγο. Όχι. Θα απαντήσω λιγάκι στο ερώτημα του κυρίου Ρούμπιχ ή μάλλον θα δώσω το λόγο προηγουμένως στην Κομισιόν. Γιατί εδώ πέρα νομίζω ότι η Κομισιόν έχει, της έχει απευθυνθεί ένα ερώτημα. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τις παρατηρήσεις που ενδεχομένω έχει να κάνει η Κομισιόν. Είναι κάπως ε, έκπληκτη που πρέπει να λάβουν το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι Τσιλίσκη. Είμαι στην ε, Διεύθυνση Α για τα φορολογικά θέματα και ασχολούμαστε και με την απλοποιημένη διαδικασία. Φυσικά έχουμε άλλους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Γι' αυτό κάναμε μια σύντομη διαβούλευση προτού πάρω τελικά εγώ το λόγο. για τα συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων. Τι κάνουμε για να εναρμονίσουμε τα τελωνία και να διευκολύνουμε τους ελέγχους. Και το δεύτερο σημείο που ετέθη ήταν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απλοποιημένη διαδικασία. Θα ήθελα να πω καταρχήν συμφωνούμε με την ε, Επιτροπή σας, <clears throat> με το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο θα Αποστείλτε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, η οποία είναι αρμόδια για την ειδική έκθεση για τα τελωνία. Αναγνωρίσουμε το ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών, περίπου 70% που είναι απλοποιημένες και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη διευκόλυνση των διαδικασιών και διευκολύνει τα μάλα τους Ευρωπαίους εμπορευόμενους και την ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς αντιμετωπίσαμε με μεγάλη σοβαρότητα την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και ξεκινήσαμε μετά από αυτήν και εντατικότερους ελέγχους στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε στο παρελθόν τέτοιους ελέγχους, αλλά είναι φανερό ότι πρέπει να κάνουμε να εντατικοποιήσουμε τις προσπαθίες μας. <clears throat> κάναμε επίσης και κάποιες συναντήσεις πληροφόρησης για τα, τους αρμόδιους των κρατών μελών. Ξεκινήσαμε και επισκέψεις ελέγχου και παρακολούθηση στα κράτη-μέλη Έχουμε κάνει 7 τέτοιες επισκέψεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία και να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας προς την Επιτροπή σας να κάνουμε επίσκεψη στα μισά κράτη-μέλη μέχρι το τέλος. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το κάνουμε βέβαια μαζί με τους συναδέλφους μας από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Η έλεγχή μας τώρα και οι συστάσεις μας για τα κάτι εστιάζονται <clears throat> στους ελέγχους πριν από το λογιστικό έλεγχο, προτού δοθεί μια έγκριση, είναι δηλαδή ουσιαστικά πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας, και θα θέλαμε <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι η ότι υπάρχει, ο, υπάρχει ότι συνάδει η αρχική διασάφηση με την οριστική διασάφηση που περιέχει τα στοιχεία για τα τελωνία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο αριθμός των πραγματικών υλικών ελέγχων δεν θα χρειαστεί να είναι τόσο υψηλό όσο αναφέρεται και φυσικά η αυτόματη ανάλυση κινδύνου είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ο στόχος μας όμως είναι όλες οι διαδικασίες ε, στα τελωνία να υπόκεινται σε μια αυτόματη ανάλυση κινδύνου. Πρέπει να πω ότι όλα αυτά που κάνουμε σε σχέση με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και σε σχέση με τις συστάσεις της δικής σας Επιτροπής, όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγχρονισμού των τελωνίων και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία και εμείς <clears throat> εντατικοποιούμε τις προσπαθίες μας και είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στο να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Κομισιόν και μέσω της ε, διαδικασίας εξυγχρονισμού των τελωνίων στην σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω για να προστατεύσουμε τη συλλογή των ιδιών Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλετε κι εσείς από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού να προσθέσετε κάτι. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι επικεφαλής της μονάδας για τους παραδοσιακούς πόρους από τη Γενική Διεύθυνση του Προϋπολογισμού και ήμουν παρόν όταν συζητήθηκε η έκθεση για, την για τις απλουστευμένες διαδικασίες. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 4 της γνωμοδότησης όπου λέγεται ότι υπάρχουν ε, πολύ υψηλού επίπεδου απώλειες από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Από έσοδο δηλαδή. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επισημανθεί ήδη από το ελεκτικό συνέδριο και έχει ενσωματωθεί μετά στην έκθεση. Επί τη βάση αυτής της εκθέσεως λοιπόν καταλήξαμε ότι η τελικά συμπεράσματα, τελικές συνέπειες αυτών των διαπιστώσεων 79 τον αριθμό με οικονομικές επιπτώσεις ε, πρέπει να κλείσουν. Κλείψαμε τις 65 εξ αυτών χωρίς οικονομικές επιπτώσεις. Διότι ε, κατετέθησαν εντωμεταξύ τα έγγραφα τα οποία δεν είχαν υποβληθεί εγκαίρως. Εν όλο λοιπόν οι, οικονομικές, οι δημοσιονομικές καλύτερα επιπτώσεις αυτών των ανομαλιών ως προς την ε, κατάθεση των εγγράφων έχει καλυφθεί. Δεν υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις. Και σας έχουμε ενημερώσει με μια προσωρινή έκθεση. Θα στείλουμε εδώ και την τελική όταν θα έχουμε τα ε, στοιχεία στο σύνολό τους. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω για τις ε, επιθεωρήσεις που κάνουμε στα κρατημέλη στους παραδοσιακούς ιδίους πόρους. Ιδιαίτερα μεριμνούμε να εξετάζουμε πώς λειτουργούν οι τελωνιακοί έλεγχοι στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα το 2009-2010 φροντίσαμε ώστε να γίνουν επιθεωρήσεις σε όλα τα συστήματα και τις στρατηγικές των κρατών μελών για τα τελωνία, σε κάθε κράτος μέλος δηλαδή, και έχουμε καταλήξει σε μια έκθεση κατόπιν αυτών των επιθεωρήσεων. Λαμβανωμένων υπόψη βεβαίω και των τελευταίων εξελίξεων στα κράτη-μέλη που συμπεριλαμβάνονται και στην έκθεση και που ακολουθούν τις παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και τις συστήσεις που γίνονται Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδίων Πόρων με τα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την παρουσίασα και στην ομάδα εργασίας για την τελωνιακή πολιτική. Την παρουσίασα στους δύο ευθύντες τελωνίων όλων των κρατών μελών. Βεβαίως, έχουμε εντοπίσει και κάποιες αδυναμίες, όπως επισημάνει και το ελεγκτικό συνέδριο στους τελωνιακούς, στα συστήματα, στα πλαίσια ελέγχου που θέτουν τα κράτη-μέλη. Αλλά εν γέννη, τα πόξη των κρατών μελών ήταν θετική και τα δύο τρίτα των ε, προβλημάτων που είχαμε εντοπίσει αντιμετωπίζονται από τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεταξύ να λάβει δράση. Και είμαι στη θέση σας για να σας δώσω τις ε, λεπτομέρειες ανά θέμα σε μια έκθεση. Για δε τις απλουστευμένες διαδικασίες είχαμε ε, ως θέμα ενός σεμιναρίου εφέτος την, ε, τις απλουστευμένες διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο όπου προσπαθήσαμε να εξετάσουμε το κατά πόσον γίνονται οι προκατακτικοί έλεγχοι ικανοποιητικά, κατά πόσον χρησιμοποιείται η αυτοματοποιημένη ανάλυση κινδύνου και πόσο συχνή είναι η δειγματοληπτική έλεγχη ή πόσο σωστή είναι η συλλογή των σχετικών στοιχείων. Ε, συμπερασματικά λοιπόν, πρέπει να πω ότι όσον αφορά το δικό μας σύστημα επιθεωρήσεων, προχωρούμε σε δράσεις συγκεκριμένες σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και φυσικά θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ε, πολύ σημαντική διάσταση ε, της ουσιαστικής λειτουργίας των τελωνίων και του συστήματος των ιδιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για αυτά τα καλά νέα που μας είπατε τουλάχιστον στο δεύτερο σκέλος της ε, παρουσίας της Επιτροπής. Ε, μέσα σε αυτά τα πολλά έγγραφα τα οποία λαμβάνουμε, ενδεχομένως να μου ξέφυγε η έκθεση στην οποία αναφέρεστε. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μου το ξαναστείλετε έτσι ώστε να τον λάβω υπόψη μου. Η κυρία Γκρέσλερ. Θα ήθελα να σκεφτούμε περισσότερο για το γενικότερο πλαίσιο εδώ και 7 χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το θέμα χωρίς να έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Μήπως δεν έχουμε αρκετές αρμοδιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πιο γρήγορα βήματα. Αν δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο προχωρούν τόσο βραδέως τα πράγματα στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτή η βραδιπορία και η χελοδρομία. Λοιπόν, πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, όπως πάντα η κυρία Κρέσλερ. Ε, ε από την πλευρά της Επιτροπής ε, μπορεί κάποιος να μας πει δύο λόγια πάνω σε αυτό, να μας πει ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, γιατί δεν προχωράει πιο γρήγορα. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, vraag ναι, βεβαίω. Ο ρόλο τη είναι τη κυρία Γκρέσσερ εδώ είναι για να κάνει δύσκολε ερωτήσει. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί, σας, μαζί σα ότι είναι δύσκολη ερώτηση. Αλλά πρέπει κανείς να καταλάβει τι εννοούμε όταν λέμε ότι η διαδικασία είναι αργή και η πρόοδος είναι αργή. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μειώνονται και οι πόροι. Από την άλλη πλευρά είναι δύσκολο να κάνουμε εκτιμήσεις. Δεν ξέρουμε ε, τι ακριβώς μας έχει διαφύγει. Ξέρουμε ότι είναι πιο αποτελεσματική η έλεγχη. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό όταν κάνουμε ελέγχους και όταν κάνουμε μετά λογιστικό έλεγχο να απαντώνται πολλά ερωτήματα και όντως απαντώνται πολλά ερωτήματα ζητήματα και όταν έχουμε υποψία ε, απάτης σε πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται η απάτη, απλώς είχαμε υποψία η οποία δεν επαληθεύθηκε. Το σημαντικό είναι να λειτουργεί το σύστημα αποτελεσματικά στα κράτη-μέλη, να κάνουν ε, και τα κράτη-μέλη δικούς τους λογιστικούς ελέγχους, ανάλυση κινδύνου. Και επίσης είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια νομική βάση, έστω και αν δεν είναι πάρα πολύ, ε, πάρα ισχυρή. Είναι ο κανονισμός 648, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται να υπάρχει ανάλυση κινδύνου στα κράτη-μέλη. Το σημαντικό λοιπόν είναι να έχουμε όλοι τις ίδιες μεθοδολογίες σε όλα τα κρατημέλη όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολύ σημαντική, έτσι πολύ θετική ε, αντιμετώπιση και αντίδραση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα θέματα αυτά με λίγο, διότι τα κράτη-μέλη ε, σε επίπεδο γενικών διευθυντών τελωνιακών αρχών ε, δήλωσαν ότι εάν η νομική βάση δεν είναι επαρκής, ε, τότε είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν παραπέρα, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα ίδιο συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους, τις μεθόδους ελέγχου και ανάλυσης κινδύνου κλπ. Υπάρχει βεβαίως και ο, ο νέος κώδικας των τελωνίων και εκεί θέλουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση και να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών. Αυτά μπορούσα να πω μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, με ενέπνευσε λίγο η ερώτηση της κυρίας Γκρέσλερ και οδηγούμε λοιπόν στο να πω ότι ίσως καλή ιδέα θα ήταν να συζητήσουμε το θέμα με τους συντονιστές. Μήπως δηλαδή για το 12-13 θα μπορούσαμε να κάνουμε μία έκθεση όσον αφορά την καλή λειτουργία των τελωνιακών αρχών, την καταπολέμηση των ανομαλιών και της απάτης. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό. Ε, να το αποφασίσουμε ε, και να αποφασίσουμε πρώτα στους συντονιστές και μετά με τη Γενική Διεύθυνση Ταξίδου και με τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού να συζητήσουμε ε, το θέμα αυτό. Θέλετε να πείτε και κάτι ακόμα? Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το περιβάλλον των τελωνίων εξελίσσεται διαρκώς, ε, διαρκώς υπάρχει απέτηση και ζήτηση για απλουστευμένες διαδικασίες, υπάρχει και μεγαλύτερος φόρτος. Τα πράγματα δεν είναι ίδια όπως ήταν 7 χρόνια πριν. Ε, επομένως οι πρακτικές εξελίσσονται και φυσικά θα πρέπει να εξελιχθεί και το σύστημα ελέγχου στα πλαίσια των νέων απλουστευμένων διαδικασιών. Πρόκειται για, μια, ε, ε, για ένα σημείο, για ένα πεδίο το οποίο εξελίσσεται διαρκώς και αυτή είναι ακριβώς και η μεγάλη πρόκληση και για μας. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε όλο και πιο στοχευμένες ε, έρευνες και θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται αποτελεσματικότερους, ε, αποτελεσματικότερες αναλύσεις κινδύνου. Ευχαριστούμε. Κανεί θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, τότε κλείνουμε αυτό το σημείο της τη διατάξης. Η προθεσμία για τις τροπολογίε είναι 12 το μεσημέρι στις 2 Σεπτεμβρίου. Και μετά θα γίνει η ψηφοφορία στην επόμενη συνεδρίασή μας. Πάμε στο σημείο 11 τώρα, με εισηγήτρια την κυρία Γκρέσλερ, σε σχέση με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Ουγγαρία. Θα γίνει αυτή η επίσκεψη. Ε, κανονικά προβλεπόταν από τις 20 ως 22 Ιουλίου να γίνει αυτή η επίσκεψη, αλλά την έχουμε αναβάλει. Έχουμε πάρει πολύ ε, τεκμηρίωσε τα θέματα αυτά και ελπίζω ότι θα είναι επωφελιστή και να μας πει η κυρία Γκρέσλε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω, εγώ θέλω να ζητήσω από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής μας να αναλάβουν αυτήν την, ε, την ηγεσία αυτής της ε, αντιπροσωπείας καταρχήν για την Ουγγαρία. Έχουμε ένα θαυμάσιο πρόγραμμα το οποίο έχουμε διαμορφώσει εγώ ήθελα στο πρόγραμμα αυτό να μάθω περισσότερο ποια σχέδια θα επισκεφθούμε. Έχουμε συμφωνήσει για την Πέμπτη το απόγευμα να πάμε στο μετρό τη Βουδαπέστης. Τρία θέματα γενικά. Το μετρό τη Βουδαπέστη που είναι το μεγαλύτερο στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχή. Μια εγκατάσταση καθαρισμού λιμάτων που είναι το μεγαλύτερο στο τομέα του περιβάλλοντος και ένα σχέδιο κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Θα συναντήσουμε και τους ε, πολιτικούς ε, της, ε, της αρχές της Ουγγαρίας. Τώρα έγινε αυτή η αναβολή γιατί είχαμε διάφορα προβλήματα. Θέλαμε να ξέρουμε καταρχήν τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη που παρουσιάζονται προβλήματα. Και το ταξίδι αυτό προβλεπόταν να γίνει 7 ε, χρόνια περίπου μετά την ένταξη της Ουγγαρίας. Θέλαμε να κάνουμε μια επικαιροποίηση των ε, γνώσεών μας σε σχέση με τα προβλήματα που έχει, που έχει η Ουγγαρία και με τη διαχείριση των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Εγώ δεν έχω διαβάσει βέβαια όλη αυτή την τεκμηρίωση, πρέπει να το πω. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να κάτσω να σπασικλήσω λιγάκι σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να πω στους ε, συναδέλφους να σκεφτούν και αυτοί, αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν μαζί μας, να σκεφτούν για όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε ήδη αναβάλει αυτή την ε, ε, αποστολή ήδη και πρέπει αυτή τη φορά να πάει πιο καλά. Θα έχουμε έξι εκπροσώπους και θα είναι και έξι από την Κομισιόν που θα μας συνοδεύουν. Ένας προς ένα θα είναι οι εκπρόσωποι της Κομισιόν μαζί μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακριβώ αυτή τη διαδρομή που είχαμε προβλέψει και θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού οι οποίοι οργάνωσαν το ταξίδι. Er, eh, Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θα ήθελαν να λάβουν το λόγο και να θέσουν ερωτήματα σε σχέση με αυτή την επίσκεψη της αντιπροσωπείας. Γι' αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκρέσλε, ότι πρέπει να, υπάρχουν επαρκής, να υπάρξει υπαρκής αριθμός ε, αντιπρόεδρων. Εγώ έχω κάνει ό,τι μπορώ κυρία Γκρέσλε. Έχω ηγηθεί δύο αντιπροσωπιών στο παρελθόν. Δίνω λοιπόν τη σκητάλη σε άλλους συναδέλφους αν θέλουν. Όχι, δεν έχετε άλλα θέματα. Επόμενο θέμα. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα γιατί δεν είναι παρόν ο εισηγητής ο κύριος Ριβελίνη. Δεν μας εμποδίζει αυτό να συζητήσουμε, αλλά... Αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό το πρόβλημα. Α, θα έρθει ο κύριος Ριβελίνη. Διακόπτουμε λοιπόν μέχρι να έρθει ο κύριος Ριβελίνη. Eh, Ήρθε ο εισηγητής μας και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της ημέρας. Όπως ξέρετε δεν θα γίνει συνεδρία των συντονιστών, αλλά αυτό το σημείο είναι σημαντικό. Έχουμε μία διαμάχη με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Είναι θέμα αρχής, όπως ξέρετε, και έχουμε αναβάλει από το Μάιο την απαλλαγή του Συμβουλίου. Ο κ. Ριβελίνη, Ριβελίνη είναι συγητής μας και μας έδωσε χθε το δεύτερο σχέδιο εκθέσεώς του, όπου μας προτείνει να αρνηθούμε και πάλι την απαλλαγή. Στο σχέδιο ψηφίσματός του μας λέει ακριβώς γιατί πρέπει να αρνηθούμε την απαλλαγή. Του δίνω λοιπόν το λόγο για να μας εξηγήσει ποιο είναι και το περιεχόμενο της έκθεσής του και ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων και ίσως δεν γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι στην, σε μια συνεδρίαση συντονιστών είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και ο κύριος Ζιρβελίνη <clears throat> θα σας το επιβεβαιώσει στην παράγραφο 4 του εγγράφου του γιατί εκεί εξηγεί ότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι αν δώσουμε μία απαλλαγή στην Κομισιόν βάσει του άρθρου 319 των συνθήκων θεωρεί το Συμβούλιο ότι έχει καλευθεί το σύνολο της διαδικασίας ε, απαλλαγής. Δηλαδή από τη στιγμή που δίνουμε απαλλαγή στην Κομισιόν είναι σαν να έχουμε δώσει και στο Συμβούλιο. Αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου, αλλά για μας είναι απόλυτα απαράδεκτη. Είναι μια καταχρηστική για μας ανάγνωση της, των συνδικών. Κύριε Ριβελίνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, και για αυτήν την ε, εισαγωγή που κάνατε, η οποία αποσαφήνισε την κατάσταση. μια απαλλαγής ε, η οποία αναμφίβολα προκαλεί μεγάλη ταραχή και προσοχή, εν πάση περιπτώσει, διότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της σημασίας που αποδίδεται στο Κοινοβούλιο τούτη τη στιγμή ε, με την έγκριση της απαλλαγής ή όχι. Ήδη είχαμε μία ε, σύντομη ανταλλαγή απόψε για την απαλλαγή και έχετε και το προσχέδιο. Επιτρέψτε μου όμως ναι, με λίγα λόγια να πω ποια είναι τα, τα ερωτήματα που εκκρεμούν ακόμα. Πέρα από αυτά που είπε ο Πρόεδρος, θα τα επαναλάβω κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε το πλαίσιο να είναι σαφές. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα ζητήματα που ακόμα βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ποια είναι αυτά που πρέπει περαιτέρω να συζητηθούν. Το Κοινοβούλιο δεν έλαβε καμία απάντηση σε σειρά ερωτημάτων που υπέβαλε σχετικά με την απαλλαγή του Συμβουλίου για την άσκηση 2009. Ερωτήματα τα οποία είχαμε υποβάλει στην πρώτη φάση της διαδικασίας. Ιδιαιτέρως είναι δύο τα σημεία τα οποία ε, δεν απαντήθηκαν ακόμα. Πρώτον, η διοίκηση του Συμβουλίου δεν δέχτηκε καμία πρόσκληση, δεν αποδέχτηκε καμία πρόσκληση να συναντήσει την αρμόδια αρχή από τη δική μας πλευρά για την απαλλαγή. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο δεν έλαβε από τη διοίκηση του Συμβουλίου τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που είχαμε ζητήσει με το ψήφισμα της 10ης Μαΐου του 2011. Φυσικά, πέρα από αυτά τα ζητήματα, προσπάθησα ιδιαίτερα ε, στην προετοιμασία του ψηφίσματος να πραγματοποιήσω μία προσεκτική νομική ανάλυση του δικαιώματος του Κοινοβουλίου να δώσει ή όχι την απαλλαγή, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις σε περίπτωση άρνησης της απαλλαγής. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν είναι ούτε παραδεκτές, ούτε αποδεκτές, ούτε λογικές οι θεωρήσεις του Συμβουλίου. Όταν λέει ότι η απαλλαγή της Κομισιόν καλύπτει και την απαλλαγή των άλλων θεσμικών οργάνων, όπως πρωτήτερα ανέφερε ο Πρόεδρος. Τέσσερις είναι οι κύριοι λόγοι για τη θέση μας αυτή. Πρώτον, στο άρθρο 319 του των συνθήκων που θα πρέπει βεβαίως να ειδωθεί υπό το φως του πεδίου εφαρμογής του, δηλαδή ε, να υφίστανται ε, ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο η εκτέλεση όλου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο 319 των συνθήκων, το Κοινοβούλιο πρέπει να ε, παίρνει ξεχωριστές αποφάσεις απαλλαγής για κάθε θεσμικό όργανο. Αρχή που το Συμβούλιο έχει σαφώς και ρητά επιβεβαιώσει ε, στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο σημείο. Η απαλλαγή δίνεται από το Κοινοβούλιο με αυτόνομο τρόπο όχι μονάχα όσον αφορά το τμήμα του προϋπολογισμού ε, που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και απέναντι στα τμήματα του προϋπολογισμού που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης άλλων θεσμικών οργάνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Τρίτον, η αυτονομία η οποία έχει επικυρωθεί από το δημοσιονομικό κανονισμό έχει επιβεβαιωθεί σε επίπεδο συνθήκων μέσω της πρόληψης του άρθρου 325 που επιβεβαιώνει την διαχειριστική αυτονομία των άλλων θεσμικών οργάνων. Βάσει όλων αυτών αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του διοικητικού προϋπολογισμού των άλλων θεσμικών οργάνων και επομένως ε, ε, έτσι όπως αναφέρεται ε, στο άρθρο 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Το τέταρτο στοιχείο είναι στοιχείο λογικής, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο μαζί με τα άλλα ε, νομικά στοιχεία. Οι αποφάσεις για απαλλαγή μπορούν να μπλοκάρουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με λίγα λόγια δηλαδή, προβληματικές όπως ε, η υπηρεσία της αστυνομίας ή της υπηρεσίας φαρμάκων θα μπορούσαν να μπλοκάρουν χωρίς ε, καμία δυνατότητα ε, έφεσης ή επανόδου τον, την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε το αίτημα του, κοινοβουλίου, του, συγγνώμη, του Συμβουλίου να προχωρήσουμε σε ένα πρωτόκολλο συνεννόησης διότι αυτό θα παραβίαζε ένα άρθρο των συνθήκων που ορίζει ότι το Συμβούλιο είναι αρχή αρμόδια για τις συστάσεις. Αλλά είναι αντίθετο και με την πρακτική που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και αντίθετο προς τις βασικές δημοκρατικές αρχές που έχουν ε, ορίσει το Κοινοβούλιο σαν ένα κεντρικό στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρώπη. Τέλος, η ίδια η ουσία και ο σκοπός της απαλλαγής είναι ότι κάθε δαπάνη που έχει προέλθει από χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να επαληθεύεται, να ελέγχεται από αυτούς που εκπροσωπούν τους, τους πολίτες, δηλαδή από το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αυτή η ε, ε, πραγματικά απλουστευμένη σκέψη. Δηλαδή ότι τα χρήματα των φορολογουμένων Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να ελέγχονται, ε, η χρήση των χρημάτων δηλαδή θα πρέπει να ελέγχεται από τους δημοκρατικά εκλεγμένους πολίτες, βουλευτές, είναι το πιο σημαντικό και απλό στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την πρώτη φάση η πρόταση ήταν να αρνηθούμε την απαλλαγή. Αλλά περαιτέρω διαδικασίες δεν ακολούθησαν. Δεν λάβαμε την απαραίτητη τεκμηρίωση και επομένως πραγματικά και ουσιαστικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην απαλλαγή. Εάν ε, αλλάξει η κατάσταση, εγώ θα είμαι ο πρώτος ως εισηγητής ο οποίος θα προτείνω τροποποίηση και εξέλιξη του κειμένου. Τελευταίο. Ενδεχομένως ε, σας έχει μοιραστεί ένα αντίγραφο με κάποιες τεχνικές ανακρίβειες ε, γιατί ε, δουλέψαμε πολύ και τις τελευταίες μέρες. Βεβαίως θα, υπάρξουν, θα υποβληθούν τροπολογίες οι οποίες θα αλλάξουν αυτές τις τεχνικές ανακρίβειες. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, να σας ευχαριστήσω γιατί όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες με στήριξαν, γιατί φυσικά το να δώσει κανείς ή να αρνηθεί την απαλλαγή είναι ε, ε, ένα, μια απόφαση με πολιτικό βάρος. Είχα την στήριξη όλων των πολιτικών ομάδων που επιβεβαιώνουν την βούληση να έχει κεντρικό ρόλο το Κοινοβούλιο και αυτό πραγματικά αποτελεί στοιχείο ικανοποίησης για μένα και κυρίως μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία της απαλλαγής με την μεγαλύτερη δύναμη που θα μπορούσε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριβελίνη για το έργο το οποίο έχετε φέρει σε πέρας. Ε, ποιος θα ήθελε τώρα να λάβει το λόγο. Κύριος Γκάιερ, κύριος Σόντεργαρτ και κυρία Γιάννης. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά κύριε Ριβελίνη και να σας συγχαρώ που μας κάνετε αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό και η δική μας πλευρά των σοσιαλδημοκρατών θεωρούμε ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε από το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση η οποία είναι μια προσπάθεια απόλυτης υπεκφύγης. Εμείς είχαμε κρατήσει μια συμφωνία με το Συμβούλιο, μια συμφωνία κυρίων και αυτό το οποίο διεκδικεί το Συμβούλιο είναι αστείο. Δεν υπάρχει καμία ρήτρα στη συμφωνία αυτή για απαλλαγή. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει αλλάξει σε σχέση με τα θέματα του προϋπολογισμού. Η Ισπανική Προεδρία είπε ότι δεν είναι αποχρόν λόγος αυτό το οποίο ε, διεκδικεί το Συμβούλιο. Και τώρα έχουμε δύο διαφορετικές ε, ε, προτάσεις οι οποίες έχουμε από το Συμβούλιο, δύο παραλλαγές η μία επιλογή του Συμβουλίου είναι αυτό το οποίο διεκδικούν ότι με την απαλλαγή της Κομισιόν απαλλάσσεται και το Συμβούλιο. Η δεύτερη είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, παροχές να, δοθεί, να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες αν και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να πράξει το ίδιο. Και εδώ το ερώτημα είναι Ποιο ελέγχει ποιον. Οι κυβερνήσει ελέγχουν τι κοινοβουλευτικέ συνελεύσει ή πρέπει να γίνεται το αντίθετο. Όταν έχουμε λοιπόν <clears throat> μια κατάσταση όπου αυτά τα οποία πράττει το Συμβούλιο δεν τη χάνουν επαρκού ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια, εμεί δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τη θέση ότι εμεί πρέπει να έχουμε την ευθύνη για την απαλλαγή και μετά από την ε, πρόοδο που έχει επιτύχει ο κύριος Σόντεργαρτ δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε. Ακόμα και αν είναι ένα συμβολικό βήμα, θα πρέπει για αυτό το λόγο να αρνηθούμε την ε, απαλλαγή του Συμβουλίου. Είναι σαφές αυτό και νομίζω ότι ε, υποστηρίζεται τον εισηγητή απόλυτα έτσι. Ο κύριος Σόντεργαρτ ως προηγούμενος εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ και να συγχαρώ τον κύριο Ριβελίνη. Κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά κύριε Ριβελίνη. Τα συμπεράσματά σας ε, είναι πολύ εύστοχα. Δεν νομίζω, Πρόεδρε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να έχουμε μια κατηγορηματική στάση εναντί του Συμβουλίου μια άκαμπτη στάση. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε ευελιξία μακροπρόθεσμα, αλλά από την άλλη θα πρέπει ε, να σημειώνεται και πρόοδο. Και αυτή την πρόοδο να την αναγνωρίζουμε, η οποία πρόοδο μπορεί να είναι μικρή μένα, αλλά σταθερή. Εδώ τώρα αυτό που σημειώνεται είναι όχι πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα κεκτημένα του παρελθόντος. Πράγμα το οποίο κρίνω όχι μόνο απαράδεκτο, αλλά ε, το βλέπω και σε μια πραγματική πρόκληση απέναντί μας. Ε, έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι σε ένα μόνο συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε και συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Ριβελίνη ε, ότι δηλαδή καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούμε να ψηφίσουμε παρά μόνο με έναν τρόπο το φθινόπωρο αλλά κύριε Ριβελίνη θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια επόμενη ευκαιρία, όταν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή. Και θα ήθελα να σας επισημάνω ένα ε, θέμα που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας τον είχε έρθει, στο σημείο 4. Υπάρχει μια αντίληψη ότι όταν δίνεται η απαλλαγή στην Επιτροπή δίνεται αυτομάτως και αν εφετέρου απαλλαγή και στο Συμβούλιο. Αυτό είναι απαράδεκτο φυσικά. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι γνώμη έχει γι' αυτό. Η εκτελεστική εξουσία τι θεωρεί ότι θα πρέπει να ισχύει. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει όταν τη δίνουμε απαλλαγή να δίνουμε αυτομάτω απαλλαγή και στο Συμβούλιο. Διότι αν ούτω φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν δεν θεωρούμε πως μας εικονοποιούν οι πληροφορίες του Συμβουλίου, τότε η μόνη λύση που μας μένει είναι να απορρίπτουμε την απαλλαγή και για την Επιτροπή. Και αν δεν το κάνουμε φέτος θα το κάνουμε του χρόνου. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση που μας μένει, η μόνη λύση που μας μένει εφόσον η Επιτροπή υποστηρίζει κατά τον, ίδιο, κατά τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο. Δηλαδή μπαίνετε εσείς στην ίδια βάρκα με το, με το Συμβούλιο και ε, ε, μοιράζεστε τη μοίρα του. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να το δούμε σήμερα και αν όχι σήμερα πάρα πολύ γρήγορα. Ερωτώ την Επιτροπή για άλλη μια φορά. Συμφωνείτε ε, ότι η απαλλαγή του, η δική σας ε, έχει την ίδια μοίρα με αυτήν του Συμβουλίου. Είναι ταυτόσημα. Ε, ο κύριος Μίλτζερ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σημειώσω τη συμφωνία μου στη θέση του κυρίου Ριβελίνη. Είναι πολύ καλό να εξασφαλιστεί ουσιαστικό έλεγχο ε, στην δράση του Συμβουλίου. Το θέμα είναι βέβαια με τι μέσα μπορούμε να πιέσουμε το Συμβούλιο να αλλάξει στάση και συμπεριφορά. Ένα μέσο να έχουμε μόνο στη θέσή μα. Να καταγγείλουμε, να εγκαταλείψουμε, να αποχωρήσουμε από την Συμφωνία Κυρίων. και να δεχθούμε ότι μπορεί ο καθένα να δίνει την απαλλαγή στον άλλο. Να δίνει και το Συμβούλιο απαλλαγή στο Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο απαλλαγή στο Συμβούλιο. Δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Μπορούμε να το δεχθούμε. Αλλά συμφωνώ και με εκείνου που είπαν ότι θα πρέπει να δώσει μια απερίφραστη απάντηση η Επιτροπή. σω να μην μπορεί να το πράξει σήμερα και ίσω θα πρέπει να ε, ζητήσουμε και μια πραγματογνωμοσύνη από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουνα στο παρελθόν εισηγητής για τα θέματα απαλλαγών, όπως και ο συνάδελφός μου από τη Δανία. Και το Συμβούλιο συμπεριφέρεται ως πυγμάχος στο ρίγκ, ο οποίος προσπαθεί να ε, αποσύσει τα χτυπήματα του αντιπάλου ή ένας, ως ένας παλαιστής ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει την, ε, την εμπλοκή. Δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Η θέση μας πρέπει να είναι σαφής. Όπως είπε η Μαργαρίτα Θάτσερ, είπε δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτή είναι μια από τις αγαπημένες της φράσεις. Εδώ δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και ο κ. Ζιβελίνη νομίζω ότι συμφωνεί με αυτό και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να πάρουμε άλλη γραμμή. Θα πρέπει να δείξουμε στο Συμβούλιο ότι μπορούμε να τους ελέγξουμε και θα τους ελέγξουμε. τουλάχιστον τη γραμματεία του Συμβουλίου. Εγώ δεν βλέπω λοιπόν άλλη οδό. Η απαλλαγή της ε, Κομισιόν δεν μπορεί να καλύπτει και το Συμβούλιο. Και αντίθετα από άλλους ε, συναδέλφους έχω μια θετική άποψη για την ε, Ουγγρική Προεδρία. Στο συγκεκριμένο όμως σημείο συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τη θέση του Ούγγρου Υπουργού. Ένας από τους προηγούμενους ομιλητές είπε και κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητής Eh, Νομίζω ότι το Συμβούλιο έχει σαμποτάρει τα, τη μικροφωνική εγκατάσταση, λέει ο πρόεδρος. Ε, ναι, ελπίζω ότι τώρα με ακούτε. Ίσως ήμουν πολύ σκληρός με το Συμβούλιο. Αλλά πιστεύω ότι πράγματι πρέπει να διαμαρτυρηθώ για αυτή τη στάση του Συμβουλίου. Εμείς πρέπει να κάνουμε το ταχύτερο δυνατό αυτά που είναι τα καθήκοντα του Κοινοβουλίου. Πρέπει να διαλέξουμε και τη σωστή τακτική και η Συμφωνία Κυρίων αυτή τη στιγμή μας εμποδίζουν ως Κοινοβούλιο να ασκήσουμε πλήρως το ρόλο μας και γι' αυτό θα πρέπει η Συμφωνία Κυρίων να καταγγελθεί, να την εγκαταλείψουμε, διότι αντιβαίνει στο πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας μιλάει για ένα εντονότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν και η επίσημη ε, επιβεβαίωση ότι έχει πιο σημαντικό ρόλο και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Πρέπει να είμαστε πραγματικά σκληροί με το Σύμβολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, όλοι και ο Πρόεδρος. Κυρία Γκρέσλε. Πολύ αστείο φαίνεται, αλλά θα πρέπει να ομολογήσω ότι μπορεί να δίνεται τώρα η απαλλαγή στην Επιτροπή, αλλά πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή ότι κινδυνεύει η απαλλαγή της προσεχής ε, χρήσης. Θα πρέπει να δούμε βέβαια αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε νομική ε, πραγματογνωμοσύνη και από τη δική μας νομική υπηρεσία, αλλά και από αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κατά πόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε πάνω σε, νέες, σε νέους όρους ε, την διαδικασία της απαλλαγής. Ας ε, τοποθετηθούν λοιπόν νομικές υπηρεσίες δυνατών. δυνατόν. Περίμενα και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ απαγοητευμένη. 32 διαφορετικές απαντήσεις από για 32 διαφορετικές ερωτήσεις που είχαμε υποβάλει. Χάθηκε το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Είναι λοιπόν λυπηρό το ότι ε, προσπαθούν με δικολαβικό τρόπο ορισμένοι να μας μπερδέψουν και να μην συζητήσουμε την ουσία των ζητημάτων. Εντάξει, ούτω ή άλλω ο δρόμο για το Λουξεμβούργο, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάντα ανοιχτό είναι. Α το συζητήσουμε, α το σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώ πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ε, επιλογή. Ούτως ή άλλως στην κρίση του ευρώ δεν πρόκειται να βοηθήσει καθόλου να δοθεί το μήνυμα πως υπάρχει εσωτερική διελκυστίνδα μεταξύ των θεσμικών οργάνων γιατί κάποια δεν θέλουν να υπαχθούν στον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Ασφαλώς κάποιοι θα χαρούν πολύ να ακούσουν τέτοια νέα. Κατά τα άλλα θα συμφωνήσω με τον εισηγητή και θα επισημάνω ότι μια και είναι εδώ το Συμβούλιο παρόνο, καλό θα είναι να δώσει τα μηνύματα που θέλει το Συμβούλιο, τα σωστά μηνύματα, στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα την υπαγάγει στον δημοσιονομικό έλεγχο των άλλων οργάνων. Αυτό θα ήθελα να δω, όντως, εάν το έχει, αν έχει αυτό το σκοπό το Συμβούλιο. για τα λοιπά, θα ήθελα να έχω απόφαση, απόφαση δικαστική. Δεν μπορώ να περιμένω ε, σε αυτή την ασάφεια πώς μπορώ άλλωστε να εξηγήσω στον ε, Ευρωπαίο πολίτη ότι δύο θεσμικά όργανα δεν μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ του και πρέπει να παραπέμψουν την υπόθεση στο δικαστήριο. Είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον δεν υπάρχει λύση, θέλω απόφαση δικαστική. για να σταματήσει αυτή η ασάφεια ως προς την απαλλαγή του Συμβουλίου η οποία διονέστε. Τι θα γίνει, θα μου κλείσετε το μικρόφωνο ή όχι. Er Οι σκοτεινές δυνάμεις νομίζω ότι επεμβαίνουν στα μικρόφωνά μας αλλά δεν θα αφήσουμε να μας επηρεάσουν. Δίνω το λόγο στην κυρία Ιάλα Σέντερ. Το πατήσε. Α. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που απουσίασα. Ακούγοντας τα, την πρόταση του κυρίου Ριβελίνη, ε, θεωρώ ότι πρέπει να λάβω το λόγο. που Θα πρέπει να ήμασταν αυστηροί και σε άλλα σημεία, αλλά εδώ σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα ήθελα να προσθέσω τα εξής δεν ξέρω πώς προβλέπετε να γίνεται σε άλλες επιτροπές, αλλά εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια παρουσία της νέας Προεδρίας ενώπιόν μας, να έρθει κάποιος από την Προεδρία ενώπιόν μας. Νομίζω ότι γενικά πρέπει η Προεδρία, όπως έχει δεσμευτεί και ενώπιον άλλων επιτροπών, να έρθει ενώπιον μας, γιατί έχει δείξει ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα, όπως παραδείγματος οι πίνακε συσχετισμού ή αντιστοίχηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε και συνάπτεται με τη διαφάνεια και την ικανότητα να έχουμε ένα πραγματικό έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως έλεγε και η κυρία Γκρέσλε προηγουμένω σε όλους τους τομεί, και αυτό περιλαμβάνει και το δημοσιονομικό έλεγχο, τον τρόπο που εφαρμόζεται λοιπόν η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη, Ίσως θα μπορούσαμε εκεί να εισαγάγουμε κάποιες τροπολο... τροποποίησεις και πιστεύω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να είναι παρούσα ενώπιόν μας η Πολωνική Προεδρία, όποιος είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποια δέσμευση από τη δική τους πλευρά για αυτό το δεύτερο τμήμα της ε, απαλλαγής του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Διαπιστώνω ότι οι συνάδελφοι συμφωνούν, ε, συγκατανεύοντας έτσι με νεύμα του κεφαλιού, για την πρόσκληση της Πολωνικής Προεδρίας και θα το κάνω. Θα δούμε, θα συμφωνήσουμε και μαζί μεταξύ μας να δούμε. Ε, μερικές φορές προτιμούν σε διάρκεια συνεδρίας συντονιστών ε, ή και κλεισμένων των θυρών. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, ε, σαν ιδέα να καλέσουμε την Πολωνική Προεδρία ναι, ξέρω κυρία Γιάλα Σέντερς ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά καμιά φορά και η Προεδρία ε, δεν δέχεται παρά μόνο και κλεισμένο των θυρών να μας ε, συναντήσει. Ε, το είχαμε και με την Ουγγρική Προεδρία. Εν πάση περιπτώσει, θα καλέσουμε σε διάλογο την Πολωνική Προεδρία δια του εκπροσώπου του. Θα προτείνουμε συνάντηση στο σύνολο της Επιτροπής μας, διαφορετικά και κλεισμένων των θυρών. Ε, λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο επαναλήφθηκε από πολλούς συναδέλφους και ε, επομένως εγώ το παραπέμπω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος μπορεί να μας ε, επιβεβαιώσει ε, ότι όταν δίνουμε την απαλλαγή στην Κομισιόν δίνουμε και στο Συμβούλιο. Ε, κοιτάξτε, όχι δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Βεβαίως λαμβάνομαι γνώση των θέσεων που έχουν διατυπωθεί και επομένως επίσημη ε, απάντηση θα λάβετε. Θα μπορούσατε να κάνετε και μια γραπτή ερώτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν έχει σημασία. Πάντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Η πρώτη μου αίσθηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει σόφρονα θέση και δεν θα ε, θελήσει να μπλεχτεί σε, αυτήν την οικογένεια, σε αυτόν τον οικογενειακό καυγά και θα προσπαθήσει να κρατήσει τη δικιά της ε, απαλλαγή ε, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα πιο επίσημο. Ε, θα σημειώσω την, ε, το, το ζήτημα το οποίο θίξατε και θα λάβετε επίσημη απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κοιτάξτε, δεν σας ζητούμε τώρα να παρεμβείτε σε, μια, σε έναν οικογενειακό καυγά, απλώς να παίξετε τον ρόλο σας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως θεματοφύλακας των συνθήκων. Δηλαδή να μας πείτε με ποιο τρόπο ε, ερμηνεύεται το άρθρο 319 των συνθήκων. Δηλαδή εάν ε, ε, θεωρείτε ότι η απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευρύνεται και προς τα άλλα θεσμικά όργανα και σας το ρωτάω γιατί είστε θεματοφύλακα των συνθήκων. Ο κύριος Γκάγερ θέλει το λόγο. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα, είναι πολύ <laughs> αστεία η θέση της Κομισιόν που λέει ότι δεν θέλει να μπλεχτεί σε αυτή τη ε, συμφωνία. Σε αυτό το θέμα μπορεί να θεωρεί η Κομισιόν ότι το Συμβούλιο έχει δίκιο και γι' αυτό δεν θέλει να εμπλακεί, αλλά σε σχέση με το θέμα αυτό του κοινοβουλευτικού ελέγχου μπορούμε να κάνουμε μία συμφωνία μεταξύ μας για το αν μπορούμε να θέσουμε μια κοινοβουλευτική ερώτηση στην Κομισιόν για το θέμα αυτό ή μπορεί να γίνει από τα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να υπογράψουν μια τέτοια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν που δεν πρόκειται μονάχα από ένα βουλευτή, αλλά είναι μια ερώτηση που τίθεται από όλου τους συντονιστές της Επιτροπής μας και θέλουν έτσι να καταδείξουν την ομοφωνία όλων στην ε, Επιτροπή μας και την ομοφωνία όλων των κοινοβουλευτικών που θέλουν να διευκρινιστεί αυτό το θέμα. Πρέπει αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί στην Ολομέλεια με την Κομισιόν. και σε σχέση με την έκθεση Ριβελίνη υπάρχει πάντα δυνατότητα να διατυπώσουμε προφορικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν για το ποια είναι η θέση της σε σχέση με, αυτή την νομική, με τους νομικούς ισχυρισμούς του Συμβουλίου. Και σε τελική λύση εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα με την έκθεση Ριβελίνη εάν προσθέσουμε και ένα ακόμα σημείο που λέει ότι η Συμφωνία Κυρίων δεν μπορεί να γίνει αναγνωριστή ως στοιχείο της, ε, της ε, απαλλαγής. Ότι δηλαδή η προφορική δήλωση της Ισπανικής Προεδρίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι νομική βάση για να θεωρείται ότι δίδεται η απαλλαγή στο Συμβούλιο. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω θα ήταν θετικό, κύριε Πρόεδρε, να θέσουμε αυτό το προφορικό ερώτημα στην Κομισιόν ή ακόμα και στη νομική ε, υπηρεσία της Κομισιόν προτού καν ξεκινήσουν οι διακοπές. Ίσως μπορούμε να ζητήσουμε και τη γνωμοδότηση της δικής μας νομικής υπηρεσίας όπως προέτεινε η κυρία Γκρέσλε. Νομίζω ότι πρέπει τα δύο θέματα να τεθούν παράλληλα και στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και την ε, νομική υπηρεσία της Κομισιόν. Κατανοώ τη θέση τη Κομισιόν, ξέρω ότι οι εκπρόσωποι της Κομισιόν δεν μπορούν εδώ να τοποθετηθούν. Αυτή η απάντηση θα προσδιορίσει σε κάποιο βαθμό και το μέλλον, το θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρέπει να το πω αυτό Εάν εσείς είσαστε έτοιμοι να αναλάβετε τα προβλήματα του Συμβουλίου, αυτό δεν θα διευκολύνει την απαλλαγή της Κομισιόν. Ήδη έχουν προβλήματα με την ε, δική σας απαλλαγή στην Κομισιόν. Φανταστείτε αν έχετε να κουβαλάτε στους ώμους σας και το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν ο πρόεδρος της Κομισιόν να τα κατανοήσει αυτό και στη συνέχεια να το διοχετεύσει και στα κατώτερα διοικητικά επίπεδα. Θα μπορούσατε λοιπόν τουλάχιστον κύριε Πρόεδρε να ζητήσετε να έχει υπάρξει μια γραμμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και την νομική υπηρεσία της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι, σε συνεργασία με τη Γραμματεία θα ακολουθήσουμε και με τον εισηγητή θα ακολουθήσουμε αυτήν την ε, γραμμή. Θα κάνουμε μια προφορική ερώτηση σε συνεννόηση όλοι. Έχουμε την παράγραφο 10 του προσχεδίου εκθέσεως ε, Ριβελίνη που μπορεί να αποτελέσει ορθή βάση εργασίας και θα μας επιτρέψει λοιπόν να ε, απευθύνομαι συγκεκριμένα ερωτήματα. Τώρα, για να υποβάλουμε κοινοβουλευτικό ερώτημα θα πρέπει να έχουμε ε, ικανό αριθμό συντονιστών και ε, μελών και επομένως μπλέκεται λίγο γραφειοκρατικά το θέμα. Στον κύριο Ριβελίνη, λοιπόν, τον εισηγητή θα δώσω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση των συναδέλφων είναι εξαιρετικά σόφρονα και νομίζω ότι η συζήτηση που κάναμε σήμερα ενισχύει ακριβώς αυτήν την κεντρική θέση που θέλουμε να παίζει το Κοινοβούλιο και την επιβεβαιώνει τη θέση αυτή. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια, να υποβάλουμε ένα ερώτημα το οποίο φυσικά εάν υπογραφεί και από τους συντονιστές θα αποκτήσει ιδιαίτερη ισχύ. Αυτό είναι σίγουρο. Και σήμερα, ίσως αυτό να είναι μια ελπίδα, ε, σήμερα ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, ε, δείξει έτσι σοφροσύνη και σοφία. Τα περιμένουμε να δούμε. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Οδηγούμεθα λοιπόν προς το τέλος της συνεδριάσεώς μας. Εύχομαι να περάσετε καλές διακοπές, αναζωογονητικές. Ελπίζω να ξεκουραστείτε και εσείς και οι συνάδελφοι και η γραμματεία και οι διερμηνείς. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους του, της Κομισιόν, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, εάν ήταν παρόντες και αν κατάλαβαν ότι θα δουλεύουμε εμείς για αυτούς το καλοκαίρι ε, και στις διακοπές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.